Σας παρακαλώ να καθίσετε. Ich erkläre die Abend. Κυρίσω την επανάληψη της Συνόδου που διακόπησε στις 10 Σεπτεμβρίου 2015. τα συνοπτικά πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν στις 19 του διατίθενται. Έχετε αντιρρήσεις, ενστάσεις από αυτόν. Παρακαλώ.